Ωραία. Παρακαλώ όσοι φεύγουν να φύγουν, ε, να αποχωρήσουν ησύχων. Ησύχως. Να συζητήσουν έξω. Δεν χρειάζεται να συζητούν εδώ. Αυτό ισχύει και για το προσωπικό των ομάδων και για όλους. Σας παρακαλώ, όσοι συζητείτε, να συζητήσετε έξω. Ώστε να χαιρετήσετε κάποιον, να τον χαιρετήσετε απ' έξω. Σημείο 11, συγγνώμη από τους συναδέλφους της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου που χρειάστηκε να περιμένουν. Αλλά συζητούσαμε ένα σημαντικό θέμα και αυτό είναι σημαντικό, θα συζητήσουμε τώρα το 11. Βοήθεια για το εμπόριο. Θέλουμε να, οι χώρες να μπορούν να προωθήσουν το εμπόριό τους για να υπάρξει εισόδημα. Ξέρουμε ότι η Επιτροπή έκανε μια ανακοίνωση για τη βοήθεια για το εμπόριο και χαίρομαι που έχουμε εμπειρογνώμονες μαζί μας. Έχουμε τον κύριο Λένοντ Μίτσι που ασκεί καθήκοντα για τον πλανήτη και την ευημερία στην Γενική Διάθεση ΔΕΒΚΟ. Λόγω της νέας συνένεσης έχουμε νέους όρους. Πλανήτης και ευημερία. Πολύ ωραία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ. Μαντλέν Τούνιγχα. Πώς προφέρετε? Τουίνιγχα. Τάουνικα. Α, ωραία. Ε, για το εμπόριο και τη δημόσια ανάπτυξη, στη βιώσιμη ανάπτυξη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και την Ιζαμπέλ Βασέ από την οργάνωση Concord. Θα ακούσουμε λοιπόν και την προοπτική των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων, σημαντικό θέμα της Επιτροπής μας και τη ΣΥΝΤΑ. Να δώσω το λόγο στον συμπρόεδρο τον κύριο Βίνκλαρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και κρυμμένοι συνάδελφοι να πω μερικά πράγματα ως ένα λάκτισμα της συζητήσεως. Λοιπόν, το θέμα που συζητούμε είναι κοινού συμφέροντος και κοινών ανησυχιών. Πήγαμε αποστολή το περασμένο καλοκαίρι για αυτό το θέμα, βοήθεια για την ανάπτυξη και είχαμε μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που υθετήθηκαν το τέλος του παρελθόντος έτους. Συνοψίζω έτσι κάποια στοιχεία για τη βοήθεια προς ανάπτυξη που ήταν μια ρηξικέλευθη πρωτοβουλία. 300 δισεκατομμύρια ταμιεύτηκαν σαν συνολικό ποσό μετά την εκκίνηση της πρωτοβουλίας 146 αναπτυσσόμενες χώρες έχουν, ε, ήταν δικαιούχες ε, αυτής της αναπτυξικής βοήθειας, κυρίως χώρες της Ασίας και Αφρικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτής από κοινού είναι η πρώτη πάροχη βοήθειας για ανάπτυξη. 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η συνολική συνεισφορά όχι μόνο μέχρι το 2014 ή περίπου 30% όλης της βοηθείας που χορηγήθηκε. Τώρα να σχολιάσω τον έγκαιρο τρόπο ή τον, την επικαιρότητα, τον επικαιρό χαρακτήρα της συζητήσεως. Ταυτόχρονα έχουμε ε, τους ε, ηγέτες, τους πολιτικούς και τους επιχειρηματικούς του Νταβός που, συνιστούν, που συζητούν μάλλον, συγγνώμη, την αυξανόμενη διαφορά και ανισότητα στον κόσμο. Λοιπόν, εάν έχει κάποια εργαλεία η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει την αυξανόμενη ανισότητα, ένα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία είναι ακριβώς η συμμετοχή ε, στην πρωτοβουλία Βοήθεια για την Ανάπτυξη. Κυρία Πρόεδρε, αν επιτρέπετε, να θέσω τρεις ερωτήσεις εκ μέρους της ΙΝΤΑ για έναρξη των συζητήσεων και μετά θα προχωρήσουμε στις παρουσιάσεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, όσον αφορά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταρχάς έχουμε τη Συμφωνία για Διευκόλυνση του Εμπορίου, αλλά δεν βλέπουμε κάποιο επιφανή ρόλο στην επικαιροποιημένη ε, στρατηγική ε, για τις διάφορες συμφωνίες για διευκόλυνση του εμπορίου. Ίδια ερώτηση μετά. Η ψηφιοποίηση και ανάγκη κάλυψης του ψηφιακού χάσματος είναι βασικό θέμα και στην Επιτροπή ΙΝΤΑ θεωρούμε ότι παρόλο που αναφέρεται στην ανακοίνωση δεν προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα. Τρίτο ερώτημα, τρίτο θέμα αφορά το ποσοστό βοηθείας που απευθύνεται ε, στις πολύ έφθαστες, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, έφθαστες χώρες. Θα ήταν όμως σωστή προσέγγιση, αλλά η βοήθεια θα πρέπει να είναι αποτελεσματική ε, χρειαζόμαστε δημιουργία δυναμικότητας. Ε, λοιπόν, αυτό πώς το προσεγγίζουμε, αυτή είναι άλλη μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους ομιλητέ, λέει η Πρόεδρος, να πω ότι αν συμφωνούν οι συγητέ για την γνωμοδότηση, δεν θα συζητήσουμε σήμερα το πρωί το σημείο 12 για την κοινή εμπορική πολιτική. Είναι γνωμοδότηση για την ίντα. Και συμφώνησαν οι συγητέ ότι θα ψηφιστεί το Φεβρουάριο. Δεν θα συζητήσουμε το σημείο 12. Αν περιμένουν κάποιοι σκιώδη από το σημείο του ενημερώνω. Έχουμε μέχρι 12 και 30 για το συγκεκριμένο σημείο και μετά θα έχουμε ε, γεύμα με την Βουλγαρική Προεδρία. Παρακαλώ τον πρώτο μιλήτη λοιπόν, αν έχει την καλοσύνη, να πάρει το λόγο. Ο κύριος Μίση από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ είναι ο που θα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τους αδέλφους Γενικής Διευθύνσης Εμπορίου να αναφερθούμε εκτενέστερα στα ερωτήματα που ετέθησαν μόλις τώρα. Έχουμε κατανομή των ρόλων σε αυτόν τον τομέα και τι να κάνουμε πιο καλά και με μεγαλύτερη σύνεση βάσει της ανακοινώσεως και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Όπως γνωρίζετε ήμασταν αρκετά επιτυχείς στην τελευταία δεκαετία. Αυτό αναφέρθηκε πρόσφατα με την Aid for Trade, τη βοήθεια για ανάπτυξη. Έχουμε 13,2 δις περίπου μέχρι το 2015 που δόθηκαν και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσης τα κράτη-μέλη έδωσαν τα χρήματα για το 1 τρίτο του Aid for Trade. Πάνω από 3.000 παρεμβάσεις έχουν εφαρμοστεί στον αντισώμενο χώρο και θετικά επηρέασαν τις χώρες εταίρους ε, και τις εμπορικές και παραγωγικές τους δυνατότητες. Αυτό σαφώς και αδαμφισβήτητα είναι ε, κάτι που γίνεται αποδεκτό που πάμε οι συζητήσεις. Και η έκθεση εποπτείας έχει αναρτηθεί στις σελίδα μας για τη βοήθεια για την ανάπτυξη και δείχνει ποικιλομορφία παρεμβάσεων. Και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων. Είναι σαφές όμως ότι τα τελευταία δέκα χρόνια το τοπίο του κόσμου έχει αλλάξει και η εκμετάλλευση της παγκοσμιοποίησης και του εμπορίου είναι κάτι πολιτικό, οικονομικό ε, και περιβαλλοντικό θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Και γίνονται συζητήσεις λοιπόν για την ανισότητα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε σε ένα παγκόσμιο πολυμερές πλαίσιο τις ανισότητες. Παρά τη βοήθεια μας, οι έφταστες χώρες παραμένουν στα περιθώρια της παγκόσμιας οικονομίας και τους λείπει παραγωγική ε, πολυμορφία. Δηλαδή, βιομηχανία στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, σύμφωνα στοιχεία του 2015, ήταν μόλις το 10%, συγκρίση με το 20% σε όλες τι αναπτυσσόμενες χώρες και το εμπορικό έλλειμμα σε αγαθά και υπηρεσίες των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών έχει ε, περίπου 10 τετραπλασιαστεί τελευταία δεκαετία από το 2006 μέχρι το 2015. 7,3 πήγε στα 104,3 εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, η βοήθεια που δίνουμε ε, δίνει συνολικά το 1 τρίτο της συνολικής βοήθειας για ανάπτυξη και επηρεάζουμε τον τρόπο με τον οποίο διατίθεται και κινητοποιείται σημαντικό κομμάτι της αναπτυξικής βοήθειας. Η βοήθεια για το εμπόριο ενεργοποιεί την βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών και έτσι μπορεί να προωθηθεί κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδος. Για να πετύχουμε τους στόχους δεν είναι θέμα μόνο αναπτυξιακής συνεργασίας, όλα τα μέσα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Και κυρίως το εμπόριο και επενδύσεις και σχετικές πολιτικές. Πώς κινητοποιούνται τα διάφορα μέσα συνεκτικά και συμπληρωματικά, αυτό καθορίζει τη συνολική μας δυνατότητα να πετύχουμε πρόοδο στο θεματολόγιο του 2030. Λοιπόν, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που υπάρχει που δεν εκμεταλλεύονται οι χώρες, να κινητοποιούμε τις συμφωνίες που έχουμε για αναπτυξιακή ενίσχυση μαζί με την, ε, τα διάφορα διαθέσιμα μέσα. Παραδείγματα. Τι θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Πρώτα απ' όλα. Να συνεχίσουμε να βοηθάμε τους αναπτυσσόμενους εταίρους μέσω εμπορικών συμφωνιών ή για ελεύθερο εμπόριο, διάφορα είδη συμφωνιών οποιασδήποτε πολυμερείς συμφωνίες γενικές, GSP+, ή οτιδήποτε όλα τα προϊόντα εκτός όπλων και να καλύπτουμε κενά ε, ανταγωνιστικότητας και να μπορέσουμε να, να βοηθήσουμε τις χώρες να καταλευθούν τα πλεονεκτήματά τους. Γεωργία, παραγωγή τροφίμων, που είναι πολύ σημαντικός τομέας για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Θέλουμε να δούμε πώς πραγματικά να δώσουμε μεγαλύτερη αξία στην παραγωγή στα χέρια του γεωργού και των ενώσεων παραγωγών. Επίσης, λοιπόν, αυτά, αυτή είναι βασική τιμή, βασικός τομέας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και κυρίως για τους νέους. Λοιπόν, όπου δεν υπάρχει με επαρκής χρήση, θέλουμε να προτείνουμε ε, λύσεις. Η βοήθεια για το εμπόριο θα βοηθήσει τις χώρες εταίρους και τους παραγωγούς να συμμορφωθούν με πρότυπα, με κανονισμούς που καθορίζουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω και έτσι τα προϊόντα του να μπορούν να εξάγονται στι δικέ μα αγορέ. Πιο συγκεκριμένα, όταν απορρίπτονται παρτίδε εξαγωγών λόγω προτύπων για λόγου υγεία, η βοήθεια για, την, ε, το εμπόριο μπορεί να βοηθήσει να εφαρμόσουν διευθυντικέ δράσει οι χώρε εταίροι. Αυτό αναφέρεται πολύ συχνά πώς η βοήθεια για το εμπόριο και τα διάφορα μέσα ανάμειξης blending instruments μπορούν να δώσουν λύσει σε περίπλοκα προβλήματα παραγωγική παραγωγικής δυναμικής, δηλαδή μέσω τεχνικής βοηθείας και μέσω συγκεκριμένων επενδύσεων. Λοιπόν, έχουμε το EIP και μέσω, μέσω τριών πυλών που θα δώσουμε και τεχνική αρρωγή για να υπάρχει ποικιλομορφία στην παραγωγή, να προωθηθεί η αξία των προϊόντων, να αυξηθεί η αξία των προϊόντων μέσω διευκολύνσεως παραγωγής και μέσω δημιουργίας μεταφορικών υποδομών. Το θέμα της ψηφιοποίησης αναφέρθηκε και όπως ξέρετε έχουμε πέντε προσεγγίσεις, πέσα μέσα, βιώσιμες ευφυείς πόλης με ψηφιακό θεματολόγιο είναι στις προτεραιότητές μας. Όπως και ο αγροτικός τομέας και οι σχετικέ επιχειρήσεις. Ψηφιακό θεματολόγιο στα πλαίσια του θεματολογίου για τις βιώσιμες πόλεις. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη ιδιαιτερότητε των λιγότερων ετοιμών χωρών και τι καταστάσει που αντιμετωπίζουν για να μπορούν να έχουν απορροφητική δυνατότητα και να ωφεληθούν οι χώρε από μεγαλύτερο ποσοστό τη βοήθεια για το εμπόριο. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα μαζί με την οικονομική ανάπτυξη. Η βοήθεια για το εμπόριο έχει ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτημα για να στηρίξει την, τις γυναίκες στο εμπόριο, να μειώσουμε τις συνέπειε αλλαγή του κλίματος και να πάμε προς πιο πράσινη οικονομία. Οι επιχειρήσεις και το εμπόριο είναι σοβαρά κίνητρα για αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη και πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε αυτά. Σαφώς αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε πραγματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων και του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών και την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι αυτοί που θα πρέπει να συμμετάσχουν. Πρέπει με αυτούς να κουβεντιάσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο κοντά στα αποτελέσματα. Οι γεωργοί, οι κοινωνικοί φορεί ε, στο ιδιωτικό τομέα ή η τοπική αυτοδίκηση, παραδείγματο χάρη. Κάτι που ξεκίνησε στο Αμπιτζάν εδώ και κάποιου μήνε, οι βιώσιμε επιχειρήσει για την Αφρική. Είναι μια διαδικασία για να κινητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα, δίνοντα του φωνή στον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντα τη θέση του ιδιωτικού τομέα και για να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα μέσω πολιτικού διαλόγου σε διάφορου τομεί. Τέλος, κλείνοντα πρέπει να κινηθούμε σε έλεγχο ποιοτικό με βάση τα αποτελέσματα για να εκμεταλλευτούμε τα μαθήματα που λάβαμε και να παρουσιάζουμε τα επιτέγματα μας. Έτσι να εκμεταλλευτούμε τη θέση που έχουμε ως ηγετικοί ε, δωρητές. Πριν το καλοκαίρι θα έχουμε την έκθεση, ε, θα επικαιροποιηθεί η έκθεση για τη βοήθεια του εμπόριου, εμπόριο, θα ε, αναφέρει περισσότερα ποιοτικά στοιχεία θα κατευθύνεται περισσότερο προς τα αποτελέσματα. Μαζί με τα κράτη-μέλη θέλουμε να συντονιστούμε. Θέλουμε να αυξήσουμε τη συλλογική δυνατότητα να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τις χώρες εταίρους, να καταπολεμήσουν τη φτώχεια και να δημιουργήσουν περισσότερες, πιο αξιοπρεπείς, καλύτερες ε, θέσεις απασχόλησης μέσω εμπορίου και μέσω επενδύσεων. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, όλοι Πρόεδρος, πάρα πολύ. Μάντλιν Τάουνιγκερ έχει το λόγο. Πάντα είναι δύσκολο το όνομά μου. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Η Γενική Διευθυνσή μας συνεργάζεται με την ΤΕΒΚΟ για το θέμα αυτό και θα πρέπει πρώτα πρώτα να συμφωνήσω με όσα μας εξήγησε ο συνάδελφος της ΤΕΒΚΟ όσον αφορά την αναθεωρημένη στρατηγική της Ένωσης για το εμπόριο. Χρειάζεται περισσότερη αποτελεσματικότητα της συνεργασίας ε, της αναπτυξιακής και της εμπορικής πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και λαμβάνεται αυτό όσον αφορά τις προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες και βέβαια η ΔΕΒΚΟ είναι η πρωτοπόρη κυρίως αρμόδια και όσον αφορά τη σχετική αναθεώρηση εμείς έχουμε εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία και βεβαίως και προσχωρήσαμε ευχαρίστως σε αυτή τη στρατηγική ούτως ώστε να έχουμε τις νέους προσανατολισμούς σε αυτή την ανακοίνωση εν του 2050 και σε όλους τους τομείς έχουμε αυτή τη νέα στρατηγική, ε, σημειώσουμε πρόοδο έτσι και έχουμε τις προτεραιότητές μας για το εμπόριο και στις εμπορικές συμφωνίες να εντάξουμε την ανάπτυξη, ε, απασχόληση, εμπλοκή της ε, κοινωνίας των πολιτών, χειραφέτηση των γυναικών, αναβάθμιση της υλοποίησης των ε, συμφωνίες συνεργασίας, μέσα για δικαιώματα, ε, εταιρική ε, κοινωνική ευθύνη. Και αυτά έχουν σχέση και με την αξιακή αλυσίδα. Και έχουμε αυτά τα παραδείγματα. Έτσι βλέπετε πώς οι προτεραιότητές μας θα ενταχθούν σε αυτήν την αναθεώρηση για να δώσουμε καινούργια όθηση στο θέμα. Επίσης να συνεργάσουμε το Aid for Trade και την εφαρμογή ε, στις ε, ε, συμφωνίες τις εμπορικές, τη βιώσιμη ανάπτυξη και περιλάβουμε και τη μερίμνα για την αλλαγή του κλίματος, για τις δομές τις κοινωνικές, αποτελεσματικότητα επομένως. Θέλουμε να πετύχουμε αυτό το σημαντικό στοιχείο του προβληματισμού μας, Τώρα και ένας άλλος τομέας που προσπαθούμε περισσότερο είναι η χειραφέτηση των γυναικών και βέβαια το, η βοήθεια μέσω του εμπορίου μπορεί να βοηθήσει και την υπόθεση των γυναικών πρόσβαση σε χρηματοδότηση, συμβουλές, ε, δικτύωση και μη περιθωριοποίηση επαγγελματική, κοινωνική και είδαμε ότι επιτεύχθηκε στο Buenos στον τον Δεκέμβριο. Είχαμε αυτή την διακήρυξη, τη δήλωση των 18 μέλων του ΠΟΕ και αυτή την κοινή δήλωση για την χειραφέτηση των γυναικών και αυτό και τώρα υλοποιούμε σε συνεργασία στενή με την ΤΕΒΚΟ. Επίσης έχουμε και άλλα παραδείγματα. Αλλά Ξέρουμε ότι πιέζει ο χρόνος. Α, και κατακλείδη να σα τονίσω και άλλο ένα στοιχείο όσον αφορά την ε, επικυροποιημένη μας ε, στρατηγική της βοήθειας με το εμπόριο. Θα πρέπει να υπάρχει πιο ε, ποιοτική παρακολούθηση των εξελίξεων με τις εκθέσεις. Αυτό είναι ένα πετυχημένο αφήγημα. Δηλαδή θα πρέπει να προβάλλουμε τις επιτυχίες μας. Θα πρέπει επίσης να ξέρουν οι εταίροι μας ποιες είναι αυτούς που προσφέρονται με την, ε, αυτή την βοήθεια του εμπορίου. Αυτά και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ λέει η πρόεδρος. Και τώρα η Ιζαμπέλ Μπρασέ του Concord θα συνεχίσει. Να μας τι γίνεται επί τόπο Αυξάνονται οι εμπορικές ροές μέσω της ενίσχυσης πιάνουν τόπο τα χρήματά μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας πω τις ε, των πολιτών με αυτό το Action Aid. Το Action Aid με έδρα το Johannesburg ανήκει στο Concord. Και για να γυρίσουμε τώρα στα πιο σημαντικά. Γιατί χρειάζεται αυτή η πολιτική ε, τη βοήθεια μέσω του εμπορίου. Γιατί η απορρίθμιση του εμπορίου δεν οδηγεί αναγκαία σε ευημερία για όλους. Και γι' αυτό και είπαμε ότι θα υπάρχει ανισότητα των εταίρων και ημών. Οπότε είπαμε ότι έτσι βοηθούμε τις αμφισόμενες χώρες ούτως ώστε να ωφεληθούν οικονομικά από την αύξηση των εμπορικών ροών. Άρα γι' αυτό θα πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο την προσέγγιση μας. Γιατί ανισότητα δεν σημαίνει μόνο ε, διαφορά πλουσίου και φτωχού. Το πρόβλημα υπάρχει και μέσα σε μια δεδομένη χώρα. Α πούμε, τι τις χώρε που τελευταία είχαν υψηλού ρυθμού ανάπτυξη. αλλά επίσης αυξήθηκε και η φτώχεια και έτσι το χάσμα της ανισότητας αυξήθηκε. Development into account in the future. Αν το λάβουμε σε αυτό υπόψη στα πλαίσια της πολιτικής βοήθειας με το εμπορίο, οπότε βλέπουμε ότι μέχρι τώρα έχει βοηθήσει αυτή η πολιτική τους ε, φτωχότερους και έχουμε την κοινή στρατηγική από το 2007 και είπαμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε καλύτερα αυτή την. Ε, πολιτική, αυτή τη στρατηγική και επίσης εξετάζουμε τις ε, εκθέσεις προόδου και βλέπουμε ότι έχουμε πάνω από 100 σελίδες για το τι έγινε το 2016. Όμως εκεί δεν περιέχονται τα στοιχεία όσο αφορά τις επιπτώσεις για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και τις επιπτώσεις για το πώς είναι το δυτικό των φτωχών. Και είπαμε όμως ότι και τα ίδια με εκείνη την ε, έκθεση διαπίστωση και Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρα χρειάζεται αυτό το mainstreaming, χρειάζεται υλοποίηση χρειάζεται να δούμε το πού πάσχει η μεθοδολογία μας και δεν μπορούσαμε να αποτυπάσουμε την πραγματικότητα. Καλά τα είπε ο ε, κύριος ε, Μίτσι. δίνεται δυσανάλογα περισσότερο βάρος στην αξιολόγηση. Αλλά χρειάζεται και ο έλεγχος και η παρακολούθηση του πώς εξελίσσονται τα πράγματα και να λαμβάνουν πάντα υπόψη αυτές τις ανισότητες. Τώρα έχουμε και άλλα θετικά στοιχεία που πρέπει να τα αναφέρουμε που έχουν σχέση με αυτή την ανακοίνωση ιδίω. Αυτή μας την ε, δέσμευση κάθε πρόγραμμα, κάθε έργο να τον αναλύουμε και από πλευρά ισότητα των φίλων και χειραφέτηση των γυναικών. Επίση, θέλουμε να βοηθήσουμε τι αξιακέ αλυσίδε και να υπάρχει τελικά προσθέμενη αξία. Πολύ σημαντικό. Ακριβώ όπω και Να μην παγιδεύονται σε μαζική παραγωγή όμορφε χώρε και έτσι να μην υπάρχει προσθεμένη αξία. Αυτό έχει σχέση βέβαια και με τις εργασιακέ συνθήκες, ε, τι αμοιβέ, την οργάνωση της εργασία ε, και αυτό επίσης πλήσει περισσότερο τι γυναίκε γιατί οι δουλειέ που κάνουν είναι χαμηλών δεξιοτήτων, χαμηλού μισθολογίου κλπ. Οπότε ανεβαίνοντα την ε, αξιακή αλυσίδα βλέπουμε ότι συναντούμε λιγότερες γυναίκες. Να, η απόδειξη των λεγόμενων. Επίσης θεωρούμε πάρα πολύ θετικό το ότι εδώ πέρα αναφέρεται κυκλική ενέργεια, πράσινη οικονομία, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά έχουν σχέση με το θύμα του 2030 και τη Συμφωνία των Παρισιών. Πολύ ωραία αυτά. Όμως, λιγότερο θετικά είναι κάποια άλλα που έχουμε επισημάνει σε αυτήν την ε, ανακοίνωση. Πολύ οικονομίστηκε αυτή η ανακοίνωση σε σχέση με το θέμα του 2004 γιατί θα, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, διακυβέρνηση, την οικονομική πρόοδο, οπότε θα πρέπει να δούμε πώς η βοήθεια της Ένωσης έχει σχέση και με τους στόχους για περιβάλλον και κοινωνία. Διάλογος, διάλογος ε, πρέπει να είναι η εποδός, θα πρέπει να είναι η λέξη κλειδί. Γιατί βλέπουμε ότι και το Κοινοβούλιο έχει διαπιστώσει όμως ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και επενδύσεις και τη σωστή συμπεριφορά. Τα έχει πει το Κοινοβούλιο και τα έχει ξαναπεί. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα ούτως ώστε ε, και σε αυτό το μέτωπο να έχουμε μια νομοθετική πλαισίωση. Άλλο ένα πρόβλημα. Ανισότητα. Η νέα συνένεση για την ανάπτυξη ρίχνει το βάρος στο πώς θα καλυφθεί η καταπολέμηση της ανισότητας για κάθε αναπτυξιακή συνεργασία. Όμως αυτά δεν τα βλέπουμε στην ανακοίνωση για τη βοήθεια μέσω του εμπορίου. Είναι απλώς μια υποσημείωση και αφορά κάποιες ευαλώτες χώρες εκεί που δεν έχει πιάσει τόπο αυτή η πολιτική για την αντιμετώπιση της ανισότητας. πρέπει να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι, να οργανωθούν η συμμετοχή των γυναικών στα επαγγελματικά. Έτσι θα στοχεύσουν αποτελεσματικά στην ανισότητα. Στο Άξιον πιστεύουμε ότι η χειραβέτηση των γυναικών εδώ πέρα αντιμετωπίζεται πολύ στενά, διότι υπάρχουν διάφοροι φραγμοί σε αυτή την υπόθεση, δηλαδή να ωφεληθούν από επενδύσεις και εμπόριο οι γυναίκες. Δεν υπάρχει αναγνώριση, δεν υπάρχει αναδιανομή των όσων κάνουν οι γυναίκες πέραν της δουλειάς. Δηλαδή τι κάνουν στο σπίτι, το νοικοκυριό, βοηθάνε τους ηλικιωμένους, βοηθάνε τους ανηλίκους, τους ασθενείς. Ε, για όλα αυτά χρειάζεται προοικοδότηση. Να είναι αναδεμητικό το αποτέλεσμα για αυτά που κάνουν οι γυναίκες. Στην ανακοίνωση λέει μόνο για κάποια μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν και θα βελτιώσουν το πεντητικό κλίμα. Ωραία αυτά. Αλλά χρειάζεται να υποστηριχθούν περισσότερο αυτέ οι υπηρεσίε που προσφέρουν Α, ναι, και κάτι τελευταίο όσον αφορά τον έλεγχο, την εποπτεία και την αξιολόγηση. Μα λέει η ανακοίνωση ότι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα κριτήρια για τις εξωτερικές επενδύσεις και τις εμπορικές συμφωνίες για την υπόθεση της ε, βοήθειας του εμπορίου. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί οι συμφωνίε ελευθερία εμπορία το παγκοσμίο, το διεθνέ εμπόριο και η ΟΥΚΤΑΝΤ κυρίω ανέδειξε το γεγονό ότι θα πρέπει και στην εσωτερική αγορά και σε περιφερειακό επίπεδο να βοηθά το εμπόριο. Αλλιώ οι χώρε γίνονται πάρα πολύ ευάλωτε γιατί εξαρτώνται υπερβολικά από τις εξαγωγέ Ε, γι' αυτό και πιστεύουμε ότι όλα αυτά που λέγεται το ελεύθερο εμπόριο ή ανακοίνωση σημαίνει ότι δεν θα ξεχάσουμε του, τους μη προνομίχους σε σχέση με το εμπόριο έχουν υπογράψει τόσε αναπτυσσόμενε χώρε με συμπορικέ συμφωνίε. Ε, θα πρέπει αυτέ οι συμφωνίε να ωφελούν τι χώρε. Να υλοποιηθούν αυτέ οι συμφωνίε. Κάθε μορφή εμπορίου. Να μην ξεχνούμε καμία τέτοια μορφή εμπορίου. Α, μάλιστα. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν, λέει ο πρόεδρο. Όλε αυτέ τι μορφέ εμπορίου να καλύψουμε. Ρίμπιχ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Οι προτάσεις αυτές ε, νομίζω είναι πολύ χρήσιμες σε όλους μας. Ξέρουμε ότι τώρα συζητάμε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, οπότε έχουμε μια δυνατότητα για να ενισχύσουμε το εμπόριο με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Διάβασα κάποιες επικεφαλίδες για τον Ντάβος, ο Αμερικανός Υπουργός Εμπορίου Wilbert Ross είπε όλες οι χώρες όλες οι άλλες ε, ανεπτυγμένες χώρες είναι θύματα του προστατευτισμού και μόνο η Αμερική είναι υπέρ του ελευθέρου, του απόλυτου ελευθέρου εμπορίου. Χρειάζεται κάποια διευκρίνηση αυτή η θέση γιατί νομίζω ότι ισχύει το αντίθετο. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να δούμε και τα πλεονεκτήματα της, της παγκοσμιοποίησης. Πολλές χώρες που ε, έπασχαν από απόλυτη ένδια δεν μπορούσαν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες των πολιτών τους και μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων, μέσω των υποδομών, μέσω της επαγγελματική κατάρτισης επέτυχαν ορισμένα πράγματα και μέσω των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Υπάρχουν τρεις ε, προτεραιότητες για μας που εκπροσωπούμε την Ένωση. Πρώτον, πρέπει να επικεντρώσουμε τις επενδύσεις μας σε τομείς που θα ωφελούν τις χώρες όπου γίνονται αυτές οι επενδύσεις, τους πολίτες. Δηλαδή να είναι όπως λέτε result driven. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να χρηματοδοτήσουμε μια εγκατάσταση καθαρισμού υδάτων που μετά δεν μπορεί να λειτουργήσει για μήνες <clears throat> επειδή δεν υπάρχουν επειδή δεν υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό <clears throat> για να την κάνει να λειτουργήσει. Πρέπει να βοηθήσουμε τις ανανεώσιμες στην Ήπεθρο γιατί η ενέργεια είναι η βάση για οποιαδήποτε άλλη παραγωγική δραστηριότητα. και ο SDG 6 καθαρό νερό είναι πολύ σημαντικός γιατί οι περισσότερες ασθένειες προκύπτουν από μολυσμένο είδωρ, νερό. Και ο δεύτερος επίσης είναι απόλυτη προτεραιότητα. η ασφάλεια και η υγεία των ζώων και των τροφίμων για να υπάρχουν και ασφαλή τρόφιμα. Και αυτά πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής μας. Και επίσης οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ούτως ώστε οι λιγότερο μένες χώρες να έχουν πρόσβαση στις αγορές και διαπιστώσαμε ότι δόθηκαν 13 δισεκατομμύρια αναπτυξιακή βοήθεια το 2015. Είναι σημαντικό ποσό και ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη σημερινή συνάντηση. Η συνεργασία για την ανάπτυξη και ο συνδυασμός της με, τη, με το εμπόριο είναι πολύ βασικό. Η συμμετοχή των μικρομεσαίων, των ε, ελευθέρων επαγγελματιών, η ανεξαρτητοποίηση των γυναικών, όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Στη Γενέβη συζητήσαμε το θέμα γυναίκες και εμπόριο και είδαμε ότι υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης και ακόμη και σε μικρές επιχειρήσεις μπορεί κανείς να επιτύχει αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι και οι εισαγωγές και οι εξαγωγές αυξάνουν την αγορεστική δύναμη, οπότε το εμπόριο είναι ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης της ένδυας και αυτό έχει να κάνει και με την κατάρτιση. Και εδώ πιστεύω ότι το θεματολόγιο ανάπτυξη τη Ντόχα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη. Είναι μια νέα δυνατότητα και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ή, συγγνώμη, Εμπορίου. Και χαίρομαι που η κοινοβουλευτική συνέλευση του ΠΟΕ στην Αργεντινή ενέκρινε ένα πολύ ενδιαφέρον ψήφισμα για να δώσει δυνατότητα και στους υπουργούς και στους διαπραγματευτέ να αλλάξουν την κατεύθυνση, να κάνουμε περισσότερα για τις χώρες αυτές Βεβαίως, η μετανάστευση έχει δύο διαστάσεις. Έχουμε το κέρδος εγκεφάλους και την απώλεια εγκεφάλων. Brain gain και brain drain. Πρέπει να βοηθήσουμε τις φτωχές χώρες να κρατήσουν το δυναμικό τους. Ιδιαίτερα στην Αφρική, όπου ζουν πάνω από ένα δις, που θα μπορούσαν να γίνουν νέοι καταναλωτές. Θα μπορούσαμε από τη μία μεριά να τους ε, πουλήσουμε δικά μας προϊόντα, αλλά να εισαγάγουμε και δικά τους προϊόντα στις αγορές μας. Γι' αυτό η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου που ξέρει πολύ καλά ότι στις ε, κεκλεισμένων των θυρών συζητήσεις υπάρχουν προστατευτικές ε, επιδιώξεις από πολλά κράτη-μέλη. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί έναντι του προστατευτισμού. Γιατί το άνοιγμα των αγορών πραγματικά καταπολεμά αποφασιστικά και αποτελεσματικά τη φτώχεια. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως θέλουμε οι ευρωπαϊκές οικονομίες να επανέλθουν στο επίπεδο των αναπτυσσομένων χώρων. Όχι, θέλουμε ευημερία για όλους. Θέλουμε όλοι να μπορούν να εργαστούν. Και συμμερίζομαι πλήρως τη γνώμη ότι πρέπει με καθαρό, διαφανή και νόμιμο τρόπο να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να βοηθήσει και η επαγγελματική κατάρτιση και η, η διάκριση των εξουσιών και η δημοκρατία πρέπει να βοηθήσουμε και τα νεα νέα κράτη-μέλη. Η Ευρώπα θα μπορούσε να αποτελεί υπόδειγμα για τις αναπτυσσόμενες χώρες για το, για πώς να αναπτυχθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Μαρία Ενά από την Επιτροπή Ίντα. Ευχαριστώ για τις διάφορες παρουσιάσεις. Όντως, πρέπει να συζητήσουμε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που χορηγούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει να κάνει με το αν βοηθάει το εμπόριο ή όχι η, ε, η βοήθεια. Για παράδειγμα, μια επένδυση για ε, ε, ε, μια εγκατάσταση καθαρισμού ύδατος που μετά δεν μπορεί να λειτουργήσει είναι θέμα αυτό. Συμφωνώ με αυτό που είπε η συνάδελφος από την κοινωνία των πολιτών. Το θέμα δεν είναι να βοηθήσουμε το εμπόριο, αλλά ποιο εμπόριο. Γιατί ξεκινάμε με την ε, αντίληψη ορισμένε φορές την εσφαλμένη ότι οποιοδήποτε εμπόριο είναι θαυμάσιο. Όχι. Στην Ευρώπη έχουμε συζητήσει πολλά θέματα για τις εμπορικές συναλλαγές. Το εμπόριο μπορεί να δημιουργήσει και θέματα, προβλήματα. Κλιματολογικά, κοινωνικά, αναδιανεμητικά και αύξηση των ανισοτήτων. Το εμπόριο μπορεί να δημιουργήσει δυσχέρειες. Άρα να βοηθήσουμε το εμπόριο, αλλά ποιου τύπου εμπόριο. Η έκθεση της UNCTAD ακριβώς τονίζει το ότι όσο περισσότερο οι ε, ασταθείς οικονομίες ε, εκτίθενται στο παγκόσμιο εμπόριο, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι ανισότητες. Κυρίως πρέπει να σας απασχολήσει η ανάπτυξη ορισμένων περιφερειών και το εμπόριο στο εσωτερικό αυτών των περιφερειών. Πριν ε, ζητήσουμε από τις χώρες αυτές να συμμορφούνται με τους φυτο-υγειονομικούς μας κανόνες, είναι σημαντικό να υπάρξουν κάποιοι εσωτερικοί κανόνες που να ισχύουν εντός της χώρας για να μπορούν να προωθήσουν το εσωτερικό τους εμπόριο. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Δεύτερον, πόσο αποτελεσματική είναι η βοήθειά μας πρέπει επιπλέον να μας, ασχολήσει, να μας απασχολήσει η αποτελεσματικότητα του εμπορίου για την ανάπτυξη. Είπατε ότι στη Γενική Διεύθυνση Trade, κυρία μου, το συζητάτε πολύ. Αλλά μόνο το συζητάτε σε αυτή τη φάση από ό,τι φαίνεται. Εμείς ως Κοινοβούλιο επίσης έχουμε υιοθετήσει πολλές απόψει για το θέμα αυτό, αλλά έχουμε πάει πολύ μακρύτερα, πολύ πέρα από το διάλογο. Για την βιώσιμη ανάπτυξη στις ε, εμπορικές συμφωνίε λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μηχανισμό κυρώσεων. Θέλουμε ένα εμπόριο που να σέβεται το περιβάλλον, να σέβεται το επίπεδο ανάπτυξης και ευημερίας της κοινωνίας. Αλλά μετά λέμε, ναι, στο κεφάλαιο αυτό το βάζουμε αυτό, αλλά αν δεν τη στηρίσετε αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα υπάρξουν κυρώσεις. Εμείς θέλουμε να υπάρξουν κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε μεγάλη δημιουργικότητα όταν ε, χρειάστηκε να αλλάξει η προστασία των επενδύσεων μέσω του ISDS, e μέσω του ISDS για να υπάρξει ένα σύστημα που θα μπορούσε να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη. Ας δείξει την ίδια δημιουργικότητα για να βρει λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, για την οποία έχουμε δεσμευτεί μέσω των Συμφωνών του Παρισίου και για την ε, προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων του πληθυσμού των χωρών αυτών. Μόνο Εάν υπάρξουν αυτές οι δύο δυνατότητες, θα βοηθήσουμε την ανάπτυξη στη χώρα. Τρίτον, λέτε, θέλουμε αναπροσανατολισμό της βοήθειας για το εμπόριο. Ποιες θα είναι οι θεμελιώδεις επιλογές όμως. Να βοηθήσουμε το εμπόριο, λέτε. Αλλά αν δημιουργεί δυσχέρειες, για παράδειγμα, για την πιστιστική αυτάρκεια και κυριαρχία των χωρών συζητάμε το Μερκοσούρ και βλέπουμε ότι στα πλαίσια του Μερκοσούρ για να παράγουν ορισμένοι γεωργοί σόγια για την εξαγωγή γιατί εμείς τρέφουμε τα ζώα μας ε, στην Ευρώπη με σόγια κυρίως από την Λατινική Αμερική για να παραχθεί λοιπόν αυτή η σόγια πρέπει να αφαιρεθεί ο πληθυσμός συγγνώμη, να αφαιρεθούν οι γέες από τον τοπικό πληθυσμό που δεν μπορεί να παράγει πλέον τρόφιμα για να φάει. Ποια θα είναι λοιπόν η προτεραιότητά σα όταν θέλετε να βοηθήσετε τι χώρε αυτέ μέσω του εμπορίου. Θα βοηθήσετε να μπορεί να τραφεί ο πληθυσμό από την ε, εγχώρια ε, παραγωγή τροφίμων ή θα βοηθήσετε τη σόγια για τη δική μας κτηνοτροφία. Όταν επενδύουμε κατόπιν στις υποδομές, λέτε να επενδύσουμε στις υποδομέ. Εάν θα μειωθεί ο αποκλεισμό, για παράδειγμα, εάν θα ενταχθεί στην οικονομία ένα δάσος για να κόψουμε τα δέντρα του για να τα εξάγουμε ή θα βοηθήσετε για παράδειγμα υγειονομικέ υποδομές που θα βοηθήσουν τον πληθυσμό και άρα θα αυξηθεί και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Τι θα δώσετε, πού θα δώσετε τα λεφτά, στις ε, υποδομές υγείας ή στις υποδομές που θα σας επιτρέψουν να εκμεταλλευτείτε ε, το πολύτιμο ξύλο κάποιων ε, δασών. Επίσης, ασχολούμεθα πολύ με τις δημόσιες επενδύσεις. Η βοήθεια για το εμπόριο είναι δημόσιες επενδύσεις. Για να βοηθήσουμε μετά την ιδιωτική ανάπτυξη. Κοιτάξτε όμως, εγώ έχω το εξή πρόβλημα. Όταν πηγαίνει κανείς στις χώρες αυτές, διαπιστώνουμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις Ας δούμε μια χώρα όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ο δημόσιος προπολογισμό είναι 6 δις. Και στην ουσία δαπανώνται 3 δις. Ο προπολογισμό του Κονγκό, που είναι μια ήπειρο ολόκληρη, είναι 3 δι ο δημόσιο προπολογισμό. Το Βέλγιο για την εκπαίδευση μόνο δαπανά 6 δι, ενώ είμαστε πολύ μικρή χώρα. Όμως ο πλούτος του Κονγκό δεν είναι ο δημόσιος προπολογισμός. Είναι οι ιδιωτικέ εταιρείε που αξιοποιούν τις πρώτες ύλες της χώρας. Τι θα κάνουμε τόσο ώστε ο πλούτος αυτός της χώρας και που παράγεται από τις πρώτες ύλε να επενδύεται στη χώρα και να μην πηγαίνει όπως γίνεται τώρα στους ε, φορολογικού παραδείσους. Θέλουμε λοιπόν μια στρατηγική βοήθεια για το εμπόριο που αφορά το 0,06% και να μην συζητήσουμε το θέμα του πώς θα βοηθήσουμε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα κέρδη τους και τα κεφάλαιά τους για να επενδύσουν στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό είναι το σημαντικό για να υπάρχει μια συνέπεια της πολιτικής μας. Οπωσδήποτε και οι ιδιωτικοί πόροι να επενδύονται στις χώρες όπου προκύπτουν να ενθαρρύνουμε τις χώρες αυτές να επενδύσουν εκεί και όχι να βγάζουν τα λεφτά τους σε φορολογικούς παραδείσους. Ευχαριστώ κύριε Σκέρν και μετά κυρία Σάντσες. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τα μηνύματα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Κοινωνίας των Πολιτών και η κυρία Μπρασέ τόνισε τη δεντολογική πτυχή όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις. Τι με ανησυχεί τα μέσα, τα ελάχιστα που έχουμε προτείνει όσον αφορά τις πολιτικές προτείνουμε. Να αυξήσουμε, θέλουμε να αυξήσουμε το εμπόριο σε μια χώρα, να έχουμε περισσότερο πλούτο και να μην υπάρχει όμως καλή κατανομή του πλούτου. Ο απολογισμός όσον αφορά τους αναψυχιακού στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι πολύ κακή στη χώρα, όμως ο παραγόμενος πλούτος είναι ανώτερος από πριν. Άρα λέμε ότι έδωσε καρπού στο εμπόριο. Και όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όσον αφορά τη μείωση των ανισοτήτων, αυτό δεν έχει συμβεί. Φταίει το εμπόριο, όχι. Ίσως λίγο, αλλά δεν είναι μόνο η αιτία του εμπόριου, αλλά οι συνδευτικές πολιτικές φταίνε, αν σε μια χώρα συγκεκριμένη. Αν έχετε δύο χώρες με την ίδια εμπορική επίδοση, στη μία ένα σύστημα φορολογικό που λειτουργεί πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, έχετε δύο παράγοντες ε, σημαντικούς ανακατανομής του πλούτου στη χώρα που βελτιώνται αποτελέσματα. Και εκεί ε, ξεκινά το πολιτικό θέμα που μας αφορά. Τι θα κάνουμε ούτω ώστε να υπερισχύει το δίκαιο των πολιτών που προστατεύονται τις χώρες. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τακτοποιήσουμε το τοίκο μα. Το ανέφερες εσύ. Ανέφερε τα δάση τα, τροπικά δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα σύστημα ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, ε, κάτι το οποίο ωφελεί τη χώρε. Στην Πολωνία έχετε μια κυβέρνηση που επιτίθεται σε πρωτογενές, σε Είναι σκάνδαλο. Σε κανένα δεν έρχεται ιδέα όμως να περιορίσει την εμπορική ελευθερία αυτού του κάτους μέλους. Εάν Εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω, στον οίκο μα δεν επιβάλλουμε την τάξη. Πώ θα επιβάλλουμε κάτι τέτοιο στην ε, Αφρική. Εγώ τι προτείνω. Μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και την ΤΕΦΚΟ να, να εξετάσουν δεχόμενέ νέα συνεργασία. Παραδείγματο χάρη, μπορούμε να έχουμε συμφωνίε που είναι πιο στεναρές όσον αφορά τη συνεργασία για την επίτευξη των στόχων ε, του, της βιώσιμης ανάπτυξης. Άρα ε, εκεί θα έχουμε ένα πόδι στις χώρες. Εμείς δεν επιβάλλουμε τώρα κάτι τέτοιο. Αποφασίζει η κυβέρνηση του Κονγκό την πολιτική που εφαρμόζει, όχι εμείς. Ε, ε λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε λόγω αυτής της αδυναμίας που έχουμε. Τελευταία σκέψη. Οι συμφωνίες συνεργασίας οικονομικής εγώ είμαι φιλελεύθερο. Εγώ είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Σαν φιλελεύθερο όμως θα ήθελα ένα σύστημα ισών ευκαιριών. Εδράζοντας τι ε, διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες εμπορικής συνεργασίας στο άρθρο 24 του ΓΚΑΤ δεν είναι αυτή η καλύτερη βάση, νομική βάση για τις διαπραγματεύσεις. Ε, ε, το είπε επανειλημμένα, διότι Εκεί αναφέρεται σε ένα εμπορικό σύστημα που συνήθιζε το 1948 και αφορούσε χώρες ε, παρομοίας ανταγωνιστικότητας λίγο πολύ. Τώρα βάζουμε στο ίδιο πλαίσιο τις χώρες που είναι υποχρεωμένες να απελευθερώσουν μεγάλο κομμάτι ε, το εμπόριό τους, ενώ υπάρχουν τεράστια κενά παραγωγικά. Όπως ε, η Νιγηρία, παραδείγματο χάρη, που μπλοκάρει τη συνεργασία ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ζητούν περισσότερη προστασία για να μπορέσει να απογειωθεί η βιομηχανία της. Και μιλώντας ότι έχουν πολύ ψηλή θνησιμότητα αυτές οι χώρες, έχουν ελάχιστα μέσα να αναπτυχθούν. Δεν κατάφερε καμία χώρα στον κόσμο να έχει ευημερία καλά κατανεμημένη στον πληθυσμό χωρίς να περάσει από μια φάση εκβιομηχάνησης να λέμε ότι τα πάντα, όλα τα κακά τα οφείλονται στο εμπόριο ή όλα τα καλά στο εμπόριο, όχι. Αλλά έχει το ρόλο του να παίξει. Το άρθρο 24 δεν είναι η καλή νομική βάση για τις διαπραγματεύσεις που σχεδόν ολοκληρώθηκαν αυτό που είναι σημαντικό νέος τρόπος συνεργασίας με τις χώρες εταίρους ούτω ώστε να έχουμε μία επιρροή στα μέσα που διαθέτουν για ανακατανομή του πλούτου εντός της χώρας Είμαστε όλοι χώρες αναπτυσσόμενες. Ε, ε υπάρχουν ε, σε αυτό το, το τομέα. Στο εμπόριο η Γερμανία είναι πρωταθλήτρια όσον αφορά την ανακατανομή όμως του πλούτου ε, είναι αναπτυσσόμενη. Ευχαριστώ. Η Λόλα Σάντσες έχει το λόγο. Λίντα, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τους προσκεκλημένους μας για όσα μας εξήγησαν. Το θέμα είναι για αυτούς τους μηχανισμούς που ότι ξεχνούμε τη διευκόλυνση των εξαγωγών. Αυτό όμως δεν ωφελεί την πλειοψηφία του κόσμου στις χώρες εκείνες. Με τις χορηγίες μας αυξάνεται το ΑΕΠ, όμως εκεί τα εισοδήματα πολύ χαμηλά και η άξιση του ΑΕΠ είναι φαινάκι ότι ωφελεί τον κόσμο. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τι γυναίκε που είναι χαμηλές αυτήν την αλυσίδα αξιών ε, και τελικά έχουν πρόσβαση ε, σε πόρους χαμηλής αξίας. Ε, ας πούμε γίνονται τηλεφωνήτριες και έχουν τις χειρότερες θέσεις εργασίας στις μεγάλες ε, επιχειρήσεις. Το θέμα είναι πώς το εμπόριο θα μπορέσει να αποδώσει, να ωφελήσει τους εταίρους μας. Πρέπει να προσπαθήσουμε ούτω ώστε οι στρατηγικοί μας και οι πολιτικές μας να έχουν επιπτώσεις θετικές στον κόσμο. Άρα θα πρέπει να μην σκεφτόμαστε μόνο το εθνικό εισόδημα. Θα πρέπει να σκεφτούμε και άλλες μεταβλητές όπως το περιβάλλον και ενισότητα των φύλων. Και η στρατηγική μας για το εμπόριο θα πρέπει να βοηθήσει ούτως ώστε να ωφεληθούν οι εταίροι για την αναδιανομή του πλούτου, για ποιοτικέ κρατικές υπηρεσίες, για υγεία και περιβάλλον. Άρα και οι υπόλοιπε πολιτικές όπως και η εμπορική να λειτουργούν όπως λες είναι και της Λισαβόνας για την ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να χαράσουμε συγκεκριμένες πολιτικές για την ισότητα των φίλων να μην είναι πάντα χαμένες οι γυναίκες. Α, και μία σκέψη σύντομη. Ήδη δύο φορές αναφέρθηκε το φόρουμ του Νταβός. Σχετικά με αυτό είπαμε ούτε είναι κάτι το θετικό, όμω πρόκειται για έναν πολυμερή οργανισμό. Εκεί συναντώνται οι πιο ισχυροί οικονομικοί παράγοντε, κρατικοί και ιδιωτικοί, και αποφασίζουν για το μέλλον του πλανήτη. Α το σκεφτούμε αυτό. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού να αποφασίζει για το μέλλον του 99% μα περί αυτού πρόκειται. Το 1% έχει πάνω το 1% του παγκοσμίου πλούτου. Και αυτό σα το λέω γιατί στη σελίδα του ίντερνετ του Νταβό λέει ότι έχουμε δεσμευτεί ούτω ώστε να βελτιώσουμε τον κόσμο. Μα, μα τόσα χρόνια ε, έχουμε το Νταβό. Έγινε καλύτερο ο κόσμο. Μα είναι δυνατόν κάποιοι άχρηστοι να είναι τόσο άχρηστοι τέλο πάντων να έχουν καταφέρει τίποτα. Μάλλον δεν το θέλουν. Το 1% κατέχει το 90%. Τίποτα θέλουν να διατηρηθεί το κατεστημένο. Ε, άρα η Επιτροπή μας θα πρέπει να μην επενεί ε, ένα τέτοιο φόρουμ σαν το Νταβός. Είναι ντροπή. Φαίνεται ότι είναι τη μόδα αυτές οι σύνοδοι κορυφής και μιλάνε για θέματα όπως είναι ισότητα, αλλά δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Δεν αρκεί απλώς να το κουβεντιάσεις το θέμα, πρέπει να κάνει κιόλα. Αυτό βλέπω συμβαίνει. Έχω κάνει δύο ερωτήσει και εγώ ίδια πριν δώσω το λόγο ξανά στου ομιλητέ μα. Πρώτα απ' όλα η διαδικασία, για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Κάνατε αυτή την ανακοίνωση. Τι γίνεται τώρα. Διότι συζητάμε στου συντονιστέ πώ αντιδρούμε σε αυτό. Θα ε, θέλατε να κάνετε και προτάσει. Τι κάνετε, έρχεται σε επαφή με τα κράτη-μέλη, συνομιλείτε με τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια διαδικασία πριν επικαιροποιηθεί η στρατηγική, υπάρχει στρατηγική, υπό ποια μορφή. Πώ μπορούμε εμεί να συμβάλλουμε. Δεύτερον, αναφέρεται σε ηθικό εμπόριο, δίκαιο εμπόριο, ευπρόσδεκτο αυτό, και καλύτερη, καλύτερη αξιολόγηση συνεπιών. Διότι δίδονται πολλά χρήματα για το βοήθεια του εμπόριο. 25% είπατε, πολλά χρήματα. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε τα αποτελέσματα. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να έχουμε κάποιε ιδέε. Τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί. Ειλικρίνεια. Εγώ Έκανα αυτά στην προηγούμενη ζωή μου, αυτά τα ε, ασχολιόμουν τα έργα. Έχει τίτλο το πρόγραμμα Βοήθεια για το εμπόριο. Αυτό το τίτλο. Βοηθά πραγματικά το εμπόριο. Υπάρχουν καλά παραδείγματα, μπορούμε να μάθουμε κάτι. Θα ήταν χρήσιμο να ξέρουμε. Και να λάβετε υπόψη αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ζητάμε από. όταν μια εταιρεία που βοηθάμε, εξετάζουμε, η εταιρεία αυτή πληρώνει του φόρου τη έχουν λογαριασμού ε, σε φορολογικούς παραδείσους, εξετάζουμε τις εταιρείε που βοηθάμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Λίγα λεπτά ο καθένα έχετε, διότι έχουμε γεύμα με τη Βουλγαρική Προεδρία συντονιστέ ε, στις 12.30. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Θα προσπαθήσω να μην δημιουργήσω πρόβλημα, μιλώντας για τον πολυμερή χαρακτήρα του ΠΟΕ και τον Ταβός η διαδικασία και τα αποτελέσματα. Είμαστε ανοιχτοί εμείς. Οι διάφορες γενικές διευθύνσεις συζητούμε περιπτώσεις και αποτελέσματα. Βοηθάει η ανάλυση του τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Να δούμε ποια συμπληρωματικότητα της δράσης των κρατών μελών. Και ίσως να, να μελετηθούν κάποιες περιπτώσεις, να δούμε τι έχει αποτελέσματα, τι δεν έχει. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό που αναφέρθηκε ε, στοιχεία που αφορούν το φύλλο ε, ε, και παρακολούθηση το μέτωπο εφαρμόζονται. Υπάρχει πρόβλημα παρακολουθήσεως των στοιχείων όσον αφορά τις, τα μεταφοπρογράμματα που εφαρμόζουμε. Δεν μπορείς να πάρεις κάποιες αποφάσεις ανευστοιχείων και τα θες επίπεδο των χωρών αυτών που βοηθάμε. Κυρίως αν μιλάμε για ανισότητες επίπεδο εισόδων νοικοκυριού και προβλήματα ανα, ανακατανομής. Αν πάτε στη δημοκρατία του Κογκό και σε κάποιες άλλες χώρες της ε, κεντρικής ε, Αφρικής είναι δύσκολο να έχει αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να δούμε τι και να υπάρχουν σε αυτά τα στοιχεία. Ποια είναι η λύση. Ένα καλό επιχειρηματικό περιβάλλον που οδηγεί σε ιδιωτικέ επενδύσεις. Δεν μπορεί να λύσει το προβλήματα ε, το εμπόριο αν εξετάσουμε περιπτώσεις και το θέμα του ασφα... της ασφάλειας εφοδιασμού σε τρόφιμα, κάτι που απασχολεί όλους ιδιαίτερος, που είμαι επικεφαλής μονάδας, που ασχολείται με θέματα τροφίμων και ασφαλούς εφοδιασμού για τα τρόφιμα. Ε, Υπεύθυνε επενδύσει για τη γεωργία και εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για μια περίοδο. Δεν μπορεί να έχει επενδύσεις η οποία δεν οδηγεί σε υπεύθυνη επένδυση για τη γεωργία και δεν λαμβάνει υπόψη κοινωνικές πτυχές, περιβαλλοντικές ε, ε, πτυχές ε, και διάφορες άλλες πτυχές. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε όσον αφορά τις επενδύσεις πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την επίγνωση της υπεύθυνη επένδυσης. Λοιπόν, είδαμε ότι υπήρξε περιθώριο στις συμφωνίες να διαπραγματευτούμε και στη γεωργία και στα τρόφιμα που παράγονται, το γεωργικό τομέα. Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται στις τοπικές αγορές περισσότερο. Η διαδικασία η αφρικανική της οικονομικής ανάπτυξης κινείται κυρίως στην τοπική αγορά. Είναι μια λύση που κινείται περισσότερο στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και η βοήθεια για το εμπόριο. Ρυθμιστικό περιβάλλον κατάλληλο, διαφανές, ισχυρός κοινωνικός διάλογος, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις για τοπική και περιφερειακή αγορά. Τίποτα δεν σταματά την Αφρικανική Ήπειρο να εμπορεύεται περιφερειακά και τοπικά. Αλλά τοπικά και περιφοριακά, αν δείτε τα στοιχεία, ε, τα στοιχεία είναι τα πιο χαμηλά, λίγο το 15% στη, στη Γεωργία. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τις τοπικές και περιφερειακές αγορές και εκεί θα πρέπει να τους δώσουμε τα αναγκαία εργαλεία και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσω πραγματικής προστήξης του υπολογισμού, με κινητοποίηση εσωτερικών πόρων, με τομιακή και η πολιτική. Αν δεν έχει το κατάλληλο περιβάλλον, ακόμα και οι ιδιωτικέ επενδύσεις δεν θα έρθουν. Και σαφώς σε κάποιες περιοχές ε, υπάρχει ε, χρειάζεται και ε, να διακινδυνεύσει κάποιε επενδύσει, αλλιώ δεν θα έρθει. Αν δεν κινητοποιήσει επενδύσει, δεν θα έρθει ιδιωτική επένδυση. Πρέπει να δούμε πώ πραγματικά μπορούμε να εξετάσουμε λεπτομέρειε σε διάφορε υποθέσει, να δούμε τι γίνεται με τι ανισότητε, αλλά να δούμε και την διοντολογική διάσταση, την περιβαλλοντική διάσταση, την κοινωνική διάσταση και πώς σχετίζονται όλα αυτά με τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το θέμα της διαδικασίας. Τι θα συμβεί. Διαδικασία. Α, μία έκθεση θα υποβληθεί τον Ιούλιο. Οπότε μέσω των γραμματιών μας μπορούμε να σε επαφή με τις διάφορες γενικές διευθύνσεις και να δούμε σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι πιο εστιασμένη η συζήτηση κάποιων περιπτώσεων και να δούμε πώς η έκθεση εν ώψη της νέας μεθοδολογίας και της αξιολόγησης που θα γίνει για τα αποτελέσματα και για την εποπτεία θα μπορεί, λέω, η έκθεση να λαμβάνει υπόψη κάποιες στοιχές που εξετέθησαν σήμερα. Πρόεδρος, θα κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό, ε, ίσως. Η Μάντλιν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, χρησιμότατα τα σχόλια. Ε, Δύο-τρία θα αναφέρω. Δεν έχω το χρόνο να κάνω περισσότερα, αλλά με τα χαρά να συνεχίσουμε κατηδίαν κάποιες συζητήσεις. Λοιπόν, η συμφωνία για τη ευκόνηση του εμπορίου, αναφέρεται κύριε Βίνκλερ, είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή που ετέθη. Δείχνει ότι δεν τονίζουμε συγκεκριμένους τομείς ε, του εμπορίου για τη βοήθεια για το εμπόριο. Άλλαξε η όλη έννοια. Όταν ξεκινήσαμε συνδέονταν πολύ με τον ΠΟΕ και τη Συμφωνία Ειδικών του Εμπορίου, όπως ομάδες χάρη ε, βοήθεια της γυναίκας κλπ. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Τώρα όμως έχουν προχωρήσει. Προσπαθούμε να απαντήσουμε στα παγκόσμια προβλήματα, την παγκοσμιοποίηση και τα διάφορα επίπεδα αξιών. Σχετικό είναι όμως αυτό που θέσατε, δεν λέω. Ένα σχόλιο ότι στιαζόμεθα πολύ στην οικονομία, είπατε. Διαφωνώ, διαφωνώ. Ήρθα από μια συνεδρίαση το πρωί με του Ολλανδού συναδέλφου του Υπουργείου Απασχόληση, του Υπουργείου Εργασία. Είναι από τα πολλά παράδειγματα που έχουμε ότι εξετάζουμε περισσότερο το πώ οι πολιτικέ θα μπορούν να είναι συμπληρωματικέ και πώ μπορούμε να συνεργαστούμε. Εγώ ε, είμαι τμήματάρχη του εμπορίου και βιώσιμη ανάπτυξη. Εγώ θα έλεγα, θα, λέω, θα έλεγα εμπόριο, οι συνάδελφοι θα πούν ε, εργασία και οι συνάδελφοί σα θα πούνε τρόφιμα και. Πρέπει να δούμε πού στεριάζουν οι ε, τα διάφορα τομεί. Δεν είναι αποκλειστικά οικονομικό θέμα αυτή η βοήθεια για το εμπόριο. Μα λένε διάφοροι άλλοι συνάδελφοι από άλλου τομεί και μα λένε τι θα κάνουμε αυτό για ανάπτυξη. Εργασία, διεθνέ γραφείο εργασία, συζητούμε πολλά πράγματα που δεν ανήκουν στο κλασικό ορισμό του εμπορίου. Έχουμε ξεπεράσει το θέμα τη εργασία και μόνο πάμε περιβάλλον, κλίμα κλπ. Δεν μπορώ να αντισταθώ, παρασχολία σε αυτό που είπε η κυρία Ρένα Ασχολούμεθα λοιπόν με αυτή τη συζήτηση των ε, λιγότερων χωρών, συζητούμε το θέμα και προσπαθούμε να δούμε τι κάνουμε. Δεν υπάρχει συμφωνία στον αφορά τις ε, στο Κοινοβούλιο ιδίω, ούτε στα κράτη-μέλη, ούτε σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Τι συζητάμε. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Παράδειγμα, αντιπροσωπείε. Βιετνάμ, παραδείγματο χάρη. Είναι μια καλή περίπτωση. Οι επικεφαλεί αντιπροσωπείων κρατών μελών συνεργάζονται άριστα. Έχουν γενική εικόνα των, όλων των προγραμμάτων, των απτυξιακών, εντοπίζουν ποιοι πολυστομητικοί ε, δεν πάνε καλά και τι θέλουν υποστήριξη. Εκεί μπορούμε να τα βελτιώσουμε και να συνεργαστούμε. Συνεργαζόμαστε με το Διεθνέ Γραφείο Εργασία είναι από τους μεγαλύτερους δωρητές, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερος δωρητής προς τα ΕΛΟ είτε για την εφαρμογή ε, του εμπορίου ή για τις διάφορες πολιτικές για τους εργαζομένους. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Θα σταματήσω εδώ. Άρα να... Για πέστε ε, λέμε θέλουμε όλοι να έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη, το είπαν και οι δύο γενικέ διευθύνσει, αλλά τι, τι κάνει η Digitrade όταν τα πήγανε στραβά διαπραγματεύσει για τη Δυτική Αφρική. Γιατί έχουμε την Ιγυρία που λέει ότι θέλω να έχουμε μια συμφωνία που να σέβεται την τοποθέτησή μας όσον αφορά την εσωτερική ανάπτυξη γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η DigiTrade λέει με την ΤΕΦΚΟ θέλουμε περιφερειακή ανάπτυξη και γι' αυτό θελήσατε να κάνετε διμερή συμφωνία με την Κάνα και την ακτή ελέφαντος του που στρέφεται κατά της περιφερειακής ανάπτυξης την, την καταστρέφει συμφωνώ να λέμε κάτι και να το κάνουμε δεν είναι να τον άλλα λέμε και αλλά να κάνουμε να έχουμε πολιτική κατά καταστροφική για την περιφερειακή ανάπτυξη. Θα πρέπει να υπάρχει συνοχή, συνέπεια. Να μην λέμε από μια μεριά ότι θέλουμε περιφερειακή ανάπτυξη και από την άλλη να έχουμε τι διμερεί συμφωνίε. Δεν ξέρω, θέλετε να απαντήσετε γρήγορα, γρήγορα. Οι διμερείς επαφές με Γκάνα και εκτήλεφαντος του αφορούσαν την προβλεψιμότητα της εμπορικής πολιτικής. Αλλιώς θα πηγαίναμε σε διακοπή των εμπορικών ροών. Αυτό θα γινόταν αν δεν ενεργούσαμε έτσι. Οπότε και εμείς θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να βοηθήσουμε την ολοκλήρωση τοπική και περιφερειακή. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και ασχέτως με τη διάσταση αυτής της περιφερειακής αναπτύξης είδατε τι γίνεται για την περιφερειακή ανάπτυξη του Cape Town και Κάιρο πόσο χρόνο πήρε. Πάρα πολύ δύσκολο 53 κατετμημένες αγορές να συντονιστούν. Ε, με το Aid for Trade αυτό προσπαθούμε. Αλλά αυτό δεν γίνεται απομονωμένα αν δεν υπάρχει σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε κάθε χώρα μια στεγανή νομοθεσία. Τι λέει το Concord, κύριε Μπρασέ. Έχετε μόνο ένα λεπτό. Θα μου αρκεί, θα μου αρκεί. Απλώ θέλω να έρθω και να συμφωνήσω με αυτά που είπατε, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη δεσμευσή μα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ανάλυση των επιπτώσεων των πρωτοβουλειών του εμπορίου και των, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίση να λάβουμε υπόψη και ε, αυτέ τι αξιολογίε των ανθρώπινων δικαιώματων. Να τα λάβουμε υπόψη και να τροποποιήσουμε κάποιε από τι ε, διατάξει των εμπορικών συμφωνίων που έχουν αρνητικέ επιπτώσει. Να, το Βιετνάμ Εκεί έχουμε τέτοιες διατάξεις. Πλήσονται οι φτωχοί από αυτή τη συμφωνία. Και να έχουμε και τα ε, μέτρα που περιχαρακώνουν την ρύθμιση Τι γίνεται με τις φορολογικές επιπτώσεις, δεν το λάβαμε αυτό υπόψη στην συμφωνία με το Βίτρα. Απ' εδώ πρέπει να σας κόψω λέει πρόεδρος και θα δούμε με τους συντονιστές τι θα κάνουμε και σας υπενθυμίζω ότι στις 2.30 ξαναρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Να μην γυρνάτε από εδώ και από εκεί. Νέος κανόν. Αυτό θα ισχύσει. 2.30. Και ευχαριστούμε τους διερμήνες. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε τους αγορητάς, την ε, DEVCO και την TRADE της Γενικής Διευθύνσης.